Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Λυπούμε που σας δόμευσα το διάλειμμα για γεύμα. Έχω και κάποιες ε, διαδικαστικές ανακοινώσεις. Στην απογευματινή μας συνεδρίαση θα παραμείνουμε ως τις 5 το απόγευμα, διότι η πρέσβυρα των κάτω χωρών είναι ασθενής. Ασθενή και ε, θα παρακαλούσε να έρθει σε συνεδρίασή μας αργότερα, τον Ιούλιο, για να δούμε μαζί της τα ίδια θέματα, αλλά στην ημερήσια διάταξη του Ιουλίου. Θα έρθει σε επαφή γραμματεία με την πρεσβεία της, των κατοχωρών. Οι διερμηνείς έχουν μία ανακοίνωση. Παρακαλώ. Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω τη εργασιακή διέναξή με τη δίκηση για τι συνθήκε εργασία μα. Σε ορισμένε καμπίνε έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διερμηνεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Αυτό ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμά του στην απεργία και συνιστά διάκριση προ τι υπόλοιπε γλώσσε. Ω εκ τούτου και σε ένδειξη ελληνική, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει σε στάσει εργασία που προβλεπόταν για τη σημερινή συνεδρίαση. Και η συνεδρία θα παραμείνουμε στην καμπίνα μέχρι τι 6.30 όπω προβλέπετε. Thank you. we start uh, of our agenda. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα συζητήσουμε εδώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Είναι χαρά μου που μπορώ να υποδεχτώ τον Διευθυντή Πιέρ Ντελσό, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή στην Γενική Διεύθυνση Grow. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστερήσεις, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και που με επιτρέπετε να σας παρουσιάσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επικεντρωθώ σε μια σειρά από βασικά στοιχεία, βασικές αρχές και μετά θα περάσω σε κάποιες λεπτομέρειες, ώστε να έχουμε και χρόνο για ρωταπαντήσεις. Το πρώτο στοιχείο, στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι ότι σε αντίθεση με το τωρινό πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, θα έχουμε ένα ενιαίο αμυντικό ταμείο για την Ευρώπη με δύο θηρίδες, την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε προπαρασκευαστικές δράσεις για την έρευνα με την EIDP αυτό που ίσως ξέρετε ότι υπερψήφισε η Επιτροπή Ήτρε το πρωί με μεγάλη πλειοψηφία. Οπότε θα έχει περατωθεί όλο αυτό μέχρι το καλοκαίρι, πριν το, τις διακοπές. Ε, η πρόταση για το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει ένα ενίο ταμείο με δύο θηρίδες. Είναι σημαντικό αυτό γιατί θέλουμε να επιμείνουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνέχεια και της έρευνας και της ανάπτυξης. Δεν θέλουμε όμως να μην συμβαδίσουν οι δύο αυτές συνιστώσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και δεν ήταν ένα πρόβλημα εύκολο να επιληθεί. Έπρεπε να το συνδυάσουμε και με τον ορίζοντα 2020, τον ορίζοντα για την Ευρώπη. Αυτό το σκέλος είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε κατά νου και κάποια άλλα σημεία στα οποία θέλω να σταθώ είναι ότι γενικώ είναι γεγονός ότι όσοι ήθελαν 10 δι για το Ταμείο θα χαρούν βλέποντας ότι έχουμε τελικά 13 δις για το Ταμείο, 4 για την έρευνα και τα υπόλοιπα για την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Είναι πιο φιλόδοξο το Ταμείο από ό,τι είχε συζητηθεί αρχικά. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ε, μια σοβαρή ένδειξη, διότι δείχνει πόση σημασία αποδίδουμε στο όλο θέμα και πόσο σημαντικό θεωρούμε αυτό το τομέα. Πρέπει να έχουμε περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των εταιριών. Αυτό το στοιχείο μπορεί να ληφθεί υπόψη. Το τρίτο στοιχείο στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι δεν επινοήσαμε εκ νέου τον τροχό. Έχουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Τώρα ολοκληρώνουμε τις συζητήσεις για το επενδυτικό εργαλείο και θεωρούμε ότι θα ήταν ανόητο να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό τώρα. Η πρόταση της Επιτροπής λοιπόν βασίζεται στο υπάρχον κείμενο, προπαρασκευαστικές δράσεις από τη μία και η IDP από την άλλη. Όμω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινό μαζί σα, είναι σαφέ ότι σε ορισμένε πτυχέ έπρεπε να απλουστεύσουμε κάποια πράγματα και να ανανεώσουμε κάποιε πτυχέ. Και πάλι όμω, επειδή δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει και επειδή θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για το μέλλον του Ταμείου να έχουμε ένα σύστημα απλούστερο, για τον λόγο αυτό το κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πόνου που μπορεί να πάρουν ήταν κάτι για το οποίο χρειαζόταν μια απλουστευμένη διαδικασία σε σχέση με το τωρινό σύστημα. Όμω, αν έχετε συγκεκριμένε ερωτήσει, παρόλα αυτά ε, είμαι στη διαθέσή σα για να απαντήσω. Δεν επινοήσαμε λοιπόν εκείνον τον τροχό, βασιστήκαμε σε όσα είχαμε και κοιτάξαμε να τα διασφαλίσουμε και στο μέλλον. Και η τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι ακόμη και αν έχουμε ένα ενίο ταμείο για την έρευνα και την ανάπτυξη, δεν θα είναι όλοι οι κανόνε ταυτόσιμοι. Θα υπάρχουν και κάποιοι ειδικοί κανόνε που θα ισχύουν για το σκέλο τη έρευνα και κάποιοι άλλοι ειδικοί για το σκέλο τη ανάπτυξη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το επίπεδο των, ε, των συμβολών που μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο περισσότερα για την έρευνα παρά για την ανάπτυξη. Η διαφορά αυτή θα παραμείνει και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ενιαίο λοιπόν το Ταμείο, αλλά όχι αναγκαστικά ένα και μόνο σύνολο κανόνων. Σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Τώρα, εάν περάσουμε λίγο περισσότερο σε λεπτομέρειες, όπως είπα, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά αποτελέσματα της διαδικασίας της συναπόφασης σε σχέση με το EIDP e και όσα συζητήσαμε ε, στο επίπεδο των προπαρασκευαστικών δράσεων. Ένα θέμα που ήταν ιδιαίτερα περίπλοκο στο πλαίσιο του Ταμείου ήταν η επιλέξιμη φορείς και τι συμμετοχή μπορεί να έχουν οι εξωευρωπαϊκές χώρες του Ταμείου. Από αυτή τη σκοπιά λάβαμε υπόψη τη λύση που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευση ε, στο προηγούμενο διάστημα και τώρα οδηγείται σε ολοκλήρωση. Είναι κάτι που μπορούν να δεχτούν όλα τα θεσμικά όργανα από ό,τι φαίνεται, εφόσον έγινε δεκτή τη διαπραγματεύσει και αυτήν θα ακολουθήσουμε. Και ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θέλω να δώσετε προσοχή είναι οι συνδεόμενες χώρες, τις χώρες ΕΦΤΑ και ΕΟΧ δυνατότητα να συμμετέχουν και αυτές στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Αυτό είναι κάπως καινούριο στοιχείο, γιατί σε σχέση με το ισχύον κείμενο για τις προπαρασκευαστικές δράσεις, το τωρινό σύστημα, η Νορβηγία ήδη συνεργάζεται, αλλά όχι για το EEIDP. Ενώ έχουμε λοιπόν ένα ενιαίο ταμείο, λάβαμε την απόφαση να ακολουθήσουμε για όλους τους δικαιούχους του ταμείου ε, την ίδια προσέγγιση. Η Νορβηγία λοιπόν μπορεί να συμμετέχει και στι δύο θηρίδε του Ταμείου. Βεβαίω αυτό το δουν περαιτέρω το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, όμω είναι μια πρόταση που θεωρούμε σημαντική. Ε, ένα άλλο στοιχείο στο οποίο μα απασχόλησε στι συζητήσει μα είναι το επίπεδο των συνεισφορών και πόσα θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα διάφορα προγράμματα. Η οροφή, το όριο που προβλέψαμε στο κείμενο βασίζεται στο τρέχον DIDP. Όμως προβλέψαμε και κάποια στοιχεία απλούστευσης, ιδίως για τις μικρομεσαίες. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να είμαστε κάπως πιο ε, διαλλακτικοί και να είναι και πιο εύληπτο το κείμενο. Αυτό προϋποθέτει και απλούστευση της διαδικασίας για τις μικρομεσαίες και τα όρια που ισχύουν για αυτέ. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε εφόσον θέλετε. Αλλά θεωρούμε ότι αποτελεί βελτίωση. Και ένα ακόμα στοιχείο που επικρίθηκε πολύ από, τις, ε, από τη βιομηχανία, από το βιομηχανικό κλάδο στην ε, τωρινή πρόταση και προσπαθήσαμε να το καλύψουμε πλέον, είναι ποιο είναι το επιλέξιμο κόστο. το κόστο θα μπορούσε να επιστραφεί από το Ταμείο. Αυτό ήταν ένα καθόλου ζήτημα, διότι η... ο βιομηχανικό κλάδο ισχυριζόταν και τα κράτη-μέλη είναι ότι υπήρχαν διαφορές σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ακόμη και αν επιστρεφόταν 1% του επιλέξιμου κόστος δεν ήταν αρκετό. Και τελικώς αυτό που πρέπει να, να καταβάλει η επιχείρηση ήταν ε, υψηλό, υψηλή τιμή, μεγάλο ποσό. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάξαμε να λάβουμε υπόψη και το έμεσο κόστος που πολλές φορές επομίζονται οι εταιρείε και επιχειρήσεις. Πάντως η άμυνα δεν είναι ένας κλασικός ε, εμπορικός κλάδος και έπρεπε να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητές του. Και εν τέλει, επειδή θέλω να σας δώσω και την ευκαιρία να θέσετε ερωτήσεις, εφόσον το επιθυμείτε, η λογική του συστήματος είναι και πάλι ίδια. Βασικά θέλουμε να ε, ενισχυθεί συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των μηχανικών τους κλάδων αλλά δεν θέλουμε συνεργασία ε, ως αυτό σκοπό. Θέλουμε τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν χάρη στο Ταμείο να οδηγήσουν στην αγορά ε, χειροπιαστού ε, απτού εξοπλισμού. Ο στόχο λοιπόν δεν είναι απλώ να κάνουμε έρευνα και ανάπτυξη στο κενό, είναι να υπάρξει συγκεκριμένο αυτό εξοπλισμό που να προσφέρει νέε δυνατότητε για τα κράτη-μέλη να είναι διαθέσιμο και να τον έχουν καλύψει με τον προπολογισμό αυτό. Ε, θα σταματήσω εδώ και θα σα δώσω το χρόνο για ερωτήσει. Thank you very much indeed, Director Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Ο κ. Ντόνζον καταρχήν. Ε, ήσασταν πολύ σαφείς. Έχω όμως μία ερώτηση. Που δεν έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο βέβαια των, της εργασίας σας, αλλά αφορά την διακυβέρνηση του Ταμείου και την κατανομή αρμοδιοτήτων. Ποιες αρμοδιότητες θα έχει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, ποιος μέσα στην Κομισιόν θα έχει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, Πώ θα διανεμηθούν αυτές στο εσωτερικό της Κομισιόν κλπ. Θα... μιλήσατε πολύ για τα ποσά, μας μιλήσατε πολύ για την επιλεξιμότητα των δαπανών κλπ. Αλλά όχι για τι αρμοδιότητε. Βέβαια, πελάτες είναι τα κράτη-μέλη, ο κλάδος της άμυνας ε, ε, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς θα, τι διακυβέρνηση θα τυχαίνει το Ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ανδρικένε. Η ερώτησή μου αφορά την σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, την Ευρωπαϊκή ε, Διευκόλυνση Ειρήνης, την ε, ε, πρωτοβουλία ε, συνδέοντας την Ευρώπη και το πρόγραμμα Horizon. Κοιτώ τα νούμερα. 13 δισεκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Άμυνας, 10,5 δισεκατομμύρια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ειρήνης, 100 δισεκατομμύρια λέει η ε, κυρία Αντρικένα για το πρόγραμμα Horizon. Πώς, αλληλώς, πώς συνδέονται αυτά μεταξύ τους και πώς αλληλοσυμπληρώνονται. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένος. Ε, πρέπει να βρίσκομαι ταυτόχρονα σε δύο-τρεις διαφορετικές συνεδριάσεις αυτές τις μέρες. Ελπίζω ότι την απάντηση στην κυρία Αντρικιένε θα μα τη δώσετε με έναν τρόπο εύληπτο ε, πώς μπορούν όλες αυτές οι πηγές χρηματοδότησης να συνδυαστούν με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Και η άλλη μου ερώτηση αφορά κάτι το οποίο είπατε και που ενδιαφέρει τον κλάδο. Το θέμα των επιλέξιμων ε, δαπανών, του επιλέξιμου κόστους. πολλές βιομηχανίες μας λένε ότι αν η επιστροφή ε, στο εθνικό επίπεδο γίνεται με διαφορετικό τρόπο από ότι ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, θα συμμετάσχουμε μεν στις, στα πιλωτικά προγράμματα κλπ. Αλλά δεν θα συμμετάσχουμε κατόπιν στο, στο πρόγραμμα ε, το 100% δεν είναι αρκετό και το 125% μπορεί να μην είναι αρκετό. Θα πρέπει να καλύπτονται όλα τα κόστη ε, των δράσεων στις οποίες θα προβαίνουν οι επιχειρήσεις ε, κατόπιν εντολής των κρατών μελών. Τώρα το αν θα είναι 100, 125, 150% των ε, επιλέξιμο, οι επιλέξιμες δαπάνες έχει πολύ μεγάλη διαφορά. δεν είναι το ίδιο. Κυρία Μόντι. Και εγώ, όπω και ο κύριος Γκάλερ, δεν κατάφερα να χωρίσω τον εαυτό μου στα δύο και να είμαι πανταχού παρούσα. Οπότε θα περιμένω να ακούσω τι απαντήσει πρώτα. Να θέσω κι εγώ μια ερώτηση. Αναφερθήκατε σε ενδεχόμενες αλλαγέ ή διευκόλυνση, χαλάρωση των διατάξεων σε ό,τι αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, μικρομεσαίες μόνο ή και τις εταιρείε ε, μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ε, θα θέλετε να μας απαντήσετε και ενδεχομένως να περάσω σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων μετά. Να ξεκινήσω στα γαλλικά να απαντήσω ότι στην ερώτηση του κ. Ντονζό σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση του συστήματο. Συμφωνώ μαζί σας. Η άμυνα είναι ένας ιδιαίτερο κλάδος όπου παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο τα κράτη-μέλη. Οπότε η Κομισιόν δεν θα υποκαταστήσει που δεν είναι τα κράτη-μέλη. Συνεπώς, τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο. Εφόσον τα ίδια τα κράτη-μέλη θα καθορίσουν το πρόγραμμα δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο. Μια επιτροπή θα συνέλθει, θα καθορίσει το πρόγραμμα εργασία και τα στοιχεία τα οποία ε, θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ε, Ταμείο. Ε, ποιος θα συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή, τα κράτη-μέλη, σε συνεργασία βέβαια με την Κομισιόν. Δεύτερον, ρόλος της Κομισιόν και ποιος θα διαχειρίζεται το Ταμείο. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ε, η διαχείριση να γίνεται άμεσα. Δηλαδή η ίδια η Κομισιόν να διαχειρίζεται το Ταμείο. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε τώρα. Θα δούμε αν αυτή θα τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υπηρεσία άμυνα δεν θα παίζει ρόλο, δεν θα παίζει κανένα ρόλο. Τα ε, σχέδια τα οποία θα αναπτυχθούν θα αγοραστούν μετά από τα κράτη-μέλη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καθοριστεί μακροπρόθεσμα η να καθοριστούν μακροπρόθεσμα οι ικανότητες ε, του, που θα αναπτύξει το Ταμείο και συνεπώς η υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Για την εσωτερική οργάνωση της Κομισιόν τώρα. Ε, δεν τολμώ να απαντήσω. Δεν θα τα αποφασίσω εγώ. Όποια όμως και αν είναι η εσωτερική οργάνωση της Κομισιόν, σίγουρα θα χρειαστούμε πρόσθετο προσωπικό, ε, εμπειρογνώμων, στους οποίους αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Ενδεχομένως θα συνεργαστούμε λοιπόν με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, είτε με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη αποσπασμένους στην Κομισιόν, είτε με ένα άλλο τρόπο, αλλά πάντως σίγουρα θα πρέπει να αναζητήσουμε εξωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες. Τώρα, αν θα δημιουργηθεί καινούργια γενική διεύθυνση ή κάτι άλλο, δεν μπορώ να το πω εγώ, δεν θα το αποφασίσω εγώ. τι, ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε εμείς. Ε, θέλουμε να στείλουμε ε, το μήνυμα ότι ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι ένας μονοπύλανς, πυλώνας. Υπάρχουν και άλλοι πυλώνες όπως αυτοί τους οποίους αναφέρατε. Ε, όλοι αυτοί όπως και η κινητικότητα, η κινητικότητα. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά μαζί είναι τεράστιο ποσό. Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα θέλουμε να εστιάσουμε στις στρατιωτικέ ικανότητες που χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ισχυρή βιομηχανία. Οπότε, πρώτο σημείο αστίασης, η αμυντική βιομηχανία. Μετά, η ε, διευκόνηση ε, έχει σχέση με Επιχειρήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε κατά κάποιο τρόπο συμπληρώνει. Τώρα, η στερεωτική κινητικότητα είναι και αυτό πολύ μεγάλο, πολύ ευρύ, διότι περιλαμβάνει εξοπλισμό. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά πρακτικά προβλήματα αδειών κλπ. προκειμένου το υλικό που υπάρχει σε ένα κράτος να μπορεί να μετακινηθεί. Ε, ο ορίζον είναι κάτι διαφορετικό. Όταν συζητούσαμε την πρόταση της Κομισιόν, αναρωτιόμασταν αν θα έπρεπε ε, το Ταμείο να τοποθετηθεί στον οριζόντα Ευρώπη. Ε, ε, ή όχι. Ε, η έρευνα, αν συγγνώμη, ε, σκεφτόμασταν αν η έρευνα θα χρηματοδοτείται από το ορίζοντα Ευρώπη ή από το Ταμείο. Τελικά αποφασίσαμε να ε, χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο. Παρ' όλα αυτά, χρειαζόμαστε μια σύνδεση μεταξύ των δύο. η έρευνα για την άμυνα θα χρηματοδοτηθεί όμως από το Ταμείο και η έρευνα για την πολιτική πτυχή θα χρηματοδοτηθεί ανάλογα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, επιλέξιμων δαπανών, ο κ. Γκάλερ έφυγε, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρονται και οι υπόλοιποι. Γνωρίζουμε ότι αυτό ανησυχεί την αμυντική βιομηχανία το κείμενο που έχουν υποβάλει δεν τους ικανοποιεί. Γιατί, τι μας λένε, μας λένε ότι εμείς χρειάζεται να πληρώσουμε υπερβολικά πολλά και μακροπρόθεσμα δεν είναι καλό για μας. Αν το κόστος συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα είναι ψηλότερο από το εθνικό κόστος, δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε. Οπότε προσπαθήσαμε να προσθέσουμε ένα άρθρο σε αυτή την πρόταση που ελπίζω ότι δείχνει πώ ακούσαμε τον κλάδο. Οπότε, ποιο σύστημα προτείνουμε. Είναι το άρθρο 16 κατά βάση της πρότασής μας. Το άρθρο 16 λέει ότι για τα έμεσα κόστη σε εσά απαντάω κύριε Γκάλερ. Για τα έμεσα κόστη έχουμε κανονικά ε, ένα ποσοστό επιστροφής 25%. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, και όπως είπατε και εσείς τις περισσότερες φορές δεν θα είναι αρκετό, τότε στη δεύτερη παράγραφο έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτό το καταποκοπήν 25% επί τη βάση των πραγματικών έμεσων, ε, του πραγματικού έμεσου κόστους. Βέβαια, χρειαζόμαστε, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ε, λογιστικές μεθόδους που θα είναι δεκτή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για, την, για τις επιχειρήσεις ε, ή θα χρησιμοποιούν το 25% αν έχουν μικρότερες δαπάνες, μικρότερες επιχειρήσεις κλπ. Οπότε εκεί δεν θα χρειαστεί, δεν θα υπάρχει πρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος, αλλά αν κάποιος, κάποια επιχείρηση θέλει περισσότερο από 25% τότε μπορεί να ε, χρηματοδοτηθεί επί τη βάση του πραγματικού έμεσου κόστους. Αυτό είναι κατά βάση το σύστημα που χρησιμοποιείται στα περισσότερα κράτη-μέλη. Σε πολλά κράτη-μέλη. Προσοχή, δεν εναρμονίζουμε τις λογιστικέ μεθόδου των κρατών μελών. Αυτό που λέμε είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εθνικές σας λογιστικέ μεθόδου υπό την προπόθεση ότι αυτέ συμμορφώνονται με την, τα κοινοτικά προαπαιτούμενα. Το συζητήσαμε επί μακρόν στις υπηρεσίες μας ε, αυτό το θέμα. Σίγουρα ο αμυντικός τομέας είναι ιδιαίτερος, έχει ιδιαιτερότητες, χρειάζονται μέτρα και διατάξεις τα οποία δεν θα χρησιμοποιούσαμε αλλού. Okay, so we... Ωραία. Τώρα έχουμε δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Κλέα, θα ήθελες το λόγο. Όχι. Ε, εγώ, εγώ λέω, ο κύριος Γκάλλορ. Για να ενημερωθούμε όλοι γενικότερα. Αν θέλουμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και να κάνουμε μια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, πρέπει να επιμείνουμε ότι πρέπει να μας αντιμετωπίσετε ισότιμα. Γιατί εμείς ως συντονιστές αποφασίσαμε ότι θέλουμε να αντιμετωπιστούμε ισότιμα και η Ήτρα θέλει να μας τα πάρει όλα. Έχουν ορίσει ήδη εισηγητή. Δεν είναι μόνο η βιομηχανική προοπτική που πρέπει να μας απασχολήσει. Εμείς ως ΕΝΤΕ βλέπουμε ποιες είναι ανάγκες των κρατών μελών, θα πρέπει να υπάρχει συναρμοδιότητα. Με βάση το άρθρο 55, νομίζω. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Σε συντονισμό με την ΑΦΕΤ. Να μας καπελώσει εντελώς η Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το σημειώνω, λέει η Πρόεδρος. Βεβαίως θα συντάξουμε μία επιστολή και θα συναντηθούμε με τον κύριο Μακάλιστα για να συζητήσουμε την περαιτέρω στρατηγική μας. Ο κύριος Τζογεύσκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσω με βάση αυτά που είπε ο κύριος Γκάλα. Δηλαδή είναι θέμα αρμοδιοτήτων μας που πρέπει να γίνονται σεβαστές. Πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε στο θέμα της ε, κινητικότητας των στρατιωτικών. Είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη, για την νομική πλευρά και για το κόστος. Αλλά υπάρχει μια διχονομία μεταξύ ΣΕΝΤΕ και ΤΡΑΝ επ' αυτού. Ποιος θα πρέπει να έχει την ε, αρμοδιότητα. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΤΡΑΝ ή πρέπει να είναι κοινή και με μας. Αναφερθήκατε σε λεπτομέρειες ε, του τομέα της άμυνας. Ξέρετε, η κινητικότητα σημαίνει χερσαίες μεταφορές, ε, θαλάσσιες μεταφορές, εναέριες μεταφορές. Και υπάρχουν και νομικά θέματα. Έχω κάποια πείρα στον τομέα αυτό. Το μεγαλύτερο εμπόριο μπορεί να είναι νομικά θέματα. Μπορεί να θέσουν προβλήματα στην κινητικότητα, ιδιαίτερα για συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένο εξοπλισμό, όχι μόνο για τους ε, στρατιωτικούς. Και νομικά εμπόδια μπορεί να ε, παρεμποδίσουν και την χρήση εξοπλισμού από άλλους, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, όταν για παράδειγμα ήταν υποπολιτική το Σαράγεβο, δεν μπορούσαν για νομικού λόγου να χρησιμοποιηθούν ουκρανικά αεροπλάνα για να βοηθήσουν. Τι θα κάνει λοιπόν το. Τι θα γίνει για να αντιμετωπίσουμε αυτές προβλε... Ε, τα προβλήματα ε, για την κινητικότητα που προκύπτουν από τα νομικά θέματα και το κόστο. Επίση, παρακαλώ την Πρόεδρο να πιέσει για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας. Έχουμε εμεί διαφορετική προσέγγιση για τα θέματα κινητικότητα των στρατιωτικών από την Τραν. Άρα πρέπει και εμεί να εμπλακούμε. Και γι' αυτό το καταποκοπήν κόστος. Πολύ καλή ιδέα. 25%. Απλουστευμένη διαδικασία. Μείωση της γραφειοκρατίας. Πολύ καλό. Αλλά πρέπει να προβλέψουμε και ένα κάποιο περιθώριο. Μπορεί τελικά να υπερβληθεί αυτό το ποσοστό και θα πρέπει να έχουμε εδώ να το καλύψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτές είναι οι ερωτήσεις του δεύτερου γύρου. Παρακαλώ απαντήστε. Καλά, δεν θα ασχοληθώ εγώ με θέματα εσωτερικής οργάνωσης του Κοινοβουλίου. Ε, αυτό είναι δικό σας θέμα. Κοιτάξτε, δεν υπευλήθησαν πολλές ερωτήσεις, αλλά ίσως αυτό να σημαίνει ακριβώς ότι δεν σας εκπλήσουν αυτά τα οποία υποβάλλουμε, ε, προτείνουμε. Όπως σας είπα, δεν, δεν επανεφευρίσκουμε τον τροχό. Τα ξέρετε. Κάτι που δεν ανέφερα στην πρώτη μου παρέμβαση. Ένα τμήμα του προπολογισμού για την έρευνα θα είναι για τις καινοτομίες παρεμπόδιση, παρεμβολής. Είναι πολύ σημαντικός τομέας. Η έρευνα πρέπει να οδηγήσει σε ανάπτυξη πρωτοτύπων, το οποίο τελικά θα γίνει ε, εξοπλισμοί που κατόπιν θα πολιθούν. Αυτή είναι η λογική. Αλλά θεωρούμε ότι ένα τμήμα του προπολογισμού πρέπει να ασχολείται με καινοτόμε και παρεμποδιστικές τεχνολογίες. Κάποιες τεχνολογίες μπορεί κάποτε να γίνουν ε, σημαντικές στον στρατιωτικό και μη στρατιωτικό τομέα. Δεν το ανέφερα αλλά τονίζω ότι πραγματικά θέλω να παραμείνει στο κείμενο, γιατί είναι πολύ σημαντικό βέβαια, θα συζητηθεί, αλλά όπως ξέρετε δεν θέλουμε να αντιγράψουμε αυτό που γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά εκεί έχουν ένα σύστημα για αυτές τις τεχνολογίες και θέλουμε κάτι παρόμοιο, όχι ενδεχόμενα τραυτώσιμο. Τώρα, να επιμείνω ιδιαίτερα λίγο περισσότερο, με βάση και την ερώτησή σας, Πρόεδρε καλύπτονται και οι mid Ξέρω ότι είναι λεπτό θέμα για κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Είναι το σύστημα που προτείνουμε και το EDIDP στα πλαίσια των προγραμμάτων PESCO. Υπάρχει ένα μπόνους όταν συμμετέχει σε προγράμματα PESCO. Και αν είσαι μια εταιρεία mid-cap, επίσης μπορούν να λάβουν μπόνους. Αλλά και για τις μικρομεσαίες προστατεύσαμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Δεν κατηγορώ κανένα. Ίσως μόνο την Κομισιόνα. Το σύστημα που προτείνουμε θα έλεγα είναι λίγο περίπλοκο. Δυσνόητο. Γι' αυτό προσπαθούμε να το απλουστεύσουμε. Καλύπτονται οι mid-cap. Δεν γίνεται καμία διάκριση κατά των mid-cap. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επανέρχομαι. η Νορβηγία που είναι μέλος ε, του ενιαίου οικονομικού χώρου μπορεί να συμμετάσχει. Όχι μόνο στις προπαρασκευαστικές αλλά σε όλες τις ενέργειες του νέου ταμείου. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Γιατί είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για άλλες τρίτες χώρες τώρα. θα εφαρμόσουν το κείμενο του EDIDP. Ο κύριος Γκάλα. Κάτι άλλο που είχα ρωτήσει και, τον Επίτροπο για τον προπολογισμό. Πριν από δύο εβδομάδες και μου είπε θα ξέρουμε την άλλη εβδομάδα. Άρα την προηγούμενη, την περασμένη εβδομάδα. Το κόστος της ΠΕΣΚΟ. Ξέρετε τι λένε οι συνθήκες. Το διοικητικό κόστος και το λειτουργικό κόστος εκτός των στρατιωτικών επιχειρήσεων πρέπει να είναι στον προπολογισμό της Ένωση. Για τα διοικητικά έξοδα είναι πάντα σαφέ, αλλά για τι λειτουργικέ δαπάνε εκτός των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα ενταχθούν όπως προβλέπει η συνθήκη στον ε, προπολογισμό σας ή δεν συμφώνησαν τα κράτη-μέλη γι' αυτό. Απάντηση. Κοιτάξτε, ο κύριος Έτινγκ τα ξέρει πολύ καλύτερα. Αλλά το ταμείο που προτείνεται δεν τα καλύπτει όλα. Δεν ξέρω την απάντηση. Αλλά θα ελέγξω και θα σας στείλω γραπτή απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι έχει αποφασίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Με συγχωρείτε, δεν θα αυτοσχεδιάσω. Θα σας στείλω ε, την ακριβή απάντηση. Πρόεδρος, άλλη μια ερώτηση. Για αυτή την ειδική μεταχείριση για την Νορβηγία. Τι σημαίνει. Ίσως ε, παρομοίως ε, να φερθούμε και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία στην οποία θα καταλήξουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, για την Νορβηγία, ίσως να υπάρχει και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της Νορβηγία και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Νορβηγία είναι εντό τη ενίας αγορά, έχει συνάψει συμφωνία με την Ένωση γιατί λοιπόν να του αποκλείσουμε. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα δεν θα αποφασίσω εγώ βεβαίω. Αλλά επειδή συμμετέχω στις συζητήσει για το Γαλιλαίο, όπως ξέρετε για το Γαλιλαίο έχει μια διάσταση ασφαλείας, έχει κάποια ασφαλή συστήματα και μία επίπτωση του Brexit είναι ότι θα εξαιρεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο από τα συστήματα αυτά. Δεν θα έχει πρόσβαση. Έχω συμμετάσχει σε συζητήσεις με εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου επ' αυτού. Και η γραμμή της Κομισιόν με έγκριση των 27 κρατών μελών και όλα αυτά είναι δημοσίως γνωστά όταν θα αποχωρήσει από την Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη χώρα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί όπως οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί και κοινοποιηθεί τώρα για τη ζήτηση για τι θα γίνει μετά το Brexit Υπάρχει αυτή η πρόταση για μια εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας. Αλλά θα γίνει. Τι θα περιέχει. Δεν θα το αποφασίσω εγώ. Είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά βεβαίως ε, θέτεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Κλέα. Δεν ήθελα να μιλήσω για τον Brexit αλλά παρακολουθούσα προσεκτικά όπως ε, φαντάζεστε. Αλλά ειλικρινά ελπίζω ότι θα υπάρξει μια στενή σχέση στον τομέα της ασφάλειας αν συμβεί το Brexit που φαίνεται να είναι το πιο πιθανό δυστυχώς αν υπάρξει Brexit τότε είναι προς το συμφέρον όλων λυπάμαι λυπάμαι που η σχέση σας με το Γαλιλαίο τελικά θα θυγεί. Α, έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά η ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι ότι θα γίνουν υποπίεση χρόνου οι διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, σε ποια υπηρεσία, σε ποια γενική διεύθυνση της Κομισιόν θα είναι η διοίκηση του Ταμείου. Ποιος θα ασχολείται. Θα μας βοηθούσε λοιπόν, εφόσον ε, μελετάμε αυτές τις προτάσεις, για να διαμορφώσουμε άποψη, να έχουμε πληρέστερη εικόνα. Ποιος θα το διοικεί το ταμείο. Γιατί ξέρετε, ανάλογα με το ποιος θα το διοικεί, αλλάζουν τα πράγματα. Έχει σημασία λοιπόν. Θα μπορούσα να σας δώσω μια πολύ απλή απάντηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενιαίος φορέας και όπου και να πάει το ίδιο είναι, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείται. Αλλά κοιτάξτε, οποιαδήποτε λύση και αν προκριθεί θα πρέπει να έχει επαρκείς πόρους και θα πρέπει να έχει μια ειδική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ασχολείται με αυτό. Πρέπει να εφαρμόσουμε όλα τα προγράμματα που θα υποβληθούν. Α συμφωνήσουμε ότι εγκριθούν τα 13 δις. Είναι πολλά λεφτά. Άρα χρειαζόμαστε και παρκές προσωπικό. Την κατάλληλη διοικητική στήριξη. Αλλά δεν θα τα αποφασίσω εγώ αυτά. Και δεν συμμετέχω στη διαμόρφωση των αυτών των θεμάτων. Ο κύριος Φλάναγκαν ήθελε να ρωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βουλευτής από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και θέλω να αναπτύξω αυτό που είπε ο κύριος ε, Γκάλερ για το δώρο της ε, μετατόπισης εδώ βλέπετε ότι λείπουν πάρα πολλά μέλη της Επιτροπής μας ενώ θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Εγώ τώρα πρέπει να σας πω ότι από αυτά που είπατε πολλά δεν μου άρεσαν. Ε, δεν θα ήθελα να έχουμε ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, αλλά τα εξηγήσατε τουλάχιστον μεγάλη σαφήνεια. Πολλές ερωτήσεις δεν τέθηκαν βέβαια γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι πολλοί το ήξεραν, όμως εγώ θέλω να μπορώ να δώσω απαντήσεις στη χώρα μου και στους ψηφοφόρους μου. Ακούω στοιχεία ότι 80% των Ευρωπαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν περισσότερη ασφάλεια και άμυνα. Εγώ ρώτησα την κυρία Μογκερίνη στο παρελθόν, που μου παρουσίασε κάποια ε, βασικά δεδομένα για την ε, ε, Ιρλανδία υποτίθεται. Αλλά μιλώντας και συζητώντας με τους ανθρώπους της χώρας μου, ξέρω ότι είμαστε ταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεν, εάν μπορούμε να μιλήσουμε για unionists ε, υπέρ της Ένωσης ε, στο πλαίσιο και στα συμφραζόμενα της Ιρλανδίας, αλλά αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα ε, ως προς την ουδετερότητα, διότι τουλάχιστον κατ' όνομα είμαστε ουδέτεροι. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ζήτημα. Ε, πολλά από αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα υποστηρίζουμε, αλλά εδώ μπορεί να αποτελέσει αυτό ένα σημείο κομβικό. Δηλαδή, αν δούμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και σκεφτούμε ότι περνάμε από την, ε, το να παράγουμε ας πούμε, τρόφιμα στο να διεξάγουμε πολέμους, αυτό δεν κρατάει την Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Θα είναι πιο εύκολο δηλαδή να μετακινούνται οι στρατοί στην Ευρώπη και μερικοί από τους δρόμους που φτιάχνονται θα διευκολύνουν. Αλλά το ερώτημα είναι, υπάρχει κανένα πόλεμο αυτή, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα υπέρ τη ειρήνη ε, όλη τη ιστορία. Και ξαφνικά αρχίζει να τίθεται το ερώτημα πώ θα περνάνε τα θωρακισμένα από την ε, Ευρώπη. Ε, τι να κάνουμε, εγώ αυτά πρέπει να πω εκ μέρους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας που εκπροσωπώ. Αν δεν σας αρέσει, τόσο το χειρότερο. Κύριε Ντεσό. Ναι. Ίσως πρωτού περάσουμε από το ότι από αντιγεωργίας, τέλος πάντων αντιπαραγωγής τροφίμων έχουμε φτάσει στην διεξαγωγή πολέμων. να σας πω ότι ασχολούμαι και με το διάστημα και τον προπολογισμό για τα διαστημικά μας προγράμματα τον έχουμε αυξήσει. Επίσης κάνουμε και πολλά που έχουν σχέση με τη Γεωργία. Έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της Ευρωπα... του Ευρωκοινοβουλίου και θα παρευρεθώ και σε άλλες όπου εξηγούμε ποια μπορεί να είναι τα ωφέλη της διαστημικής πολιτικής για τη Γεωργία. Γεωργία ακριβία και ούτω καθεξής. Πολλά μπορεί να προκύψουν από το διάστημα. Όμως και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει περισσότερα κονδύλια για το διάστημα, που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για πολλέ πολιτικέ, ε, μεταξύ των οποίων η γεωργία, όχι μόνο, και η θαλάσσια και ούτω καθεξή. Αλλά παραμένω ένας απλός υπάλληλο της Επιτροπής, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για το δικό σας ερώτημα πολιτικός, όμως, χωρίς να μπορώ να την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την σκοπιά ενός πολίτη, Υποθέτω ότι όλοι πριν μερικά χρόνια ζούσαμε μια ήσυχη και χαρούμενη ζωή μέχρι να συμβούν ας πούμε οι επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει ακριβώς πόλεμος, αλλά δεν μπορούμε να γνώουμε ότι δεν ζούμε πια σε έναν κόσμο εντελώ ασφαλή. Και θα πάψω εδώ, διότι τα υπόλοιπα δεν είναι δική μου δουλειά να τα σχολιάσω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον ε, αναπληρωτή διευθυντή Ντελσό για αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε ακόμα τρία σημεία στην ημέρα διάταξη. Παρακαλώ, χειροκροτήστε μαζί μου. Thank you. debriefing. Colleagues, please be seated. Next point is in association. Παρακαλώ καθίστε. Επόμενο σημείο αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Βρίσκομαι σε θέση κάπως δυσάρεστη, διότι δεν είναι εδώ το κυρία Καηλίου, το κύριο Κίρτσος. Και δεν μπορούσαν να έρθουν στις Βρυξέλλες σήμερα, οπότε θα παρουσιάσω εγώ τα συμπεράσματα από την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Την αιρεινή σύνοδο της κοινοβουλευτικής ε, συνέλευσης. Πέντε βουλευτές ε, συμμετείχαν και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο νόημα ότι ήταν εκεί και η κυρία Καηλή και ο κύριος Κίρτσος, επίσης ο κύριος Μπούζεκ, πρόεδρος της Επιτροπής Ήτρε, η κυρία Νορίτα Νικολάη που συμμετέχει στις Επιτροπές ΕΝΤΑ και ΑΦΕΤ και εγώ η ίδια. Συμμετείχαμε σε μια ποικιλία σε όλες ε, τις επιτροπές που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Συμμετείχαμε στις συζητήσεις και το αποτέλεσμα της Συνόδου ήταν συνολικά να εκπονηθούν 16 εκθέσεις που υποβλήθηκαν και ψηφίστηκαν όπως επίσης και αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης γιατί ήταν στο πρώτο στάδιο της εκπόνησης του σε μερικές περιπτώσεις. Τα θέματα ήταν μεταξύ άλλων η ασφάλεια της περιοχής για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη με την απειλή εξανατολής που ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες σταθήκαμε στην κατάσταση που επικράτησε στα κράτη της Βαλτικής, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μια από τις εκθέσεις επικεντρώθηκε στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου περιοχή με ανάλογε δυσκολίε όπω η δική μα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κύβερνο ασφάλεια, στην συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως σε αυτόν τον ε, τομέα που αποτελεί ιδιαίτερο παράδειγμα Επίσης μας απασχόλησε η ανάπτυξη δεσμών με το ΝΑΤΟ, διότι θυμάμαι να γίνεται κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Ολομέλειά της, χωρίς την συμπερίληψη τέτοιων θεμάτων, για πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν επηρεάσει την κατάρτιση της ατζέντα του, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Συζητήθηκε στρατιωτική κινητικότητα και παρουσιάσεις για θέματα ασφαλείας από τη σκοπιά των χωρών υποδοχής έγιναν ε, για την ε, συγκεκριμένη περίπτωση της Πολωνίας με είπα τους αξιωματούχους όπως ο πρόεδρος της Πολωνίας ε, οι πρόεδροι των δύο σωμάτων της Βουλής ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών ο Υπουργός Άμυνας Βεβαίω. το τελευταίο μέρος της Συνόδου Λομέλειας αφοσιώθηκε στις συζητήσεις, αφιερώθηκε μάλλον στις συζητήσεις κατόπιν πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιάνν Στόλτενμπερκ στα θέματα αυτά. Ήταν δική του η ομιλία με μια ευρεία συζήτηση με συμμετοχή και δική μας, δική μου, της κυρίας Καϊλή Θέσαμε ερωτήσεις, υπήρξε διάλογος και βεβαίως μας συνόδευσαν και μέλη της γραμματείας. Επικεφαλής της γραμματείας νομίζω αυτά είχα να πω. Παρακαλώ. Λίγο δύσκολο για μένα την ίδια, διότι εγώ εκπροσωπώ ούτως ή άλλως σε ένα βαθμό την Επιτροπή ΣΕΝΤ σε αυτή την αντιπροσωπεία, αλλά προσπάθησα να είμαι αντικειμενική και ακριβής. Ίσως αμέσως να περάσω στην επόμενη απενημέρωση ad hoc αντιπροσωπεία στην Γεωργία. 7 ε, έως 10 Μαΐου. ανοιξιάτικη επίσκεψη ανταλλάξαμε, ε, μάλλον συναντηθήκαμε με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, μετά είχαμε μια σειρά από συναντήσεις και επαφές με τους ανώτερους αξιωματούχους της χώρας, της Γεωργίας, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Συμφιλίωσης, καθώς και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Συναντήσαμε τον πρόεδρο της Γεωργιανής Βουλής και προέδρους των ε, πλέον ε, οικείων σε δικά μας θέματα κοινοβουλευτικών επιτροπών. με μια διακομματική σύνθεση πολλές φορές. Προσεκλήθησαν όλοι. Νομίζω υπήρχε καλή εκπροσώπηση πέρα από κάποιες αρχικές ε, παρατηρήσεις που είχαν γίνει. Και όπως και στο παρελθόν, από προηγούμενη αντιπροσωπεία της ΕΝΤ ε, και επίσκεψη στη Γεωργία, Είχαμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων, ακούσαμε κάποιες ε, παρουσιάσεις για να ενημερωθούμε, είχαμε συζήτηση με εκπροσώπους του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης του ΝΑΤΟ στη Γεωργία και κατόπιν της νορβηγικής πρωτοβουλίας να ε, διευκολύνουμε τέτοιου είδους προγράμματα χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα αυτό ακριβώς από το ΝΑΤΟ, τα μέλη του ΝΑΤΟ και στην ομιλία μου προς, το, ε, προς τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική συνέλευση ε, όταν μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και αποτίμησα το έργο αυτού του κέντρου εκπαίδευσης ε, τοποθετήθηκα θετικά. Είναι σημαντικό το κέντρο γιατί διευκολύνει την Γεωργία στην προσπάθειά της να εξυγχρονίσει ε, τον στρατό της, τις ειδικές της δυνάμεις. Την επόμενη ημέρα, τρίτη ημέρα παρουσίας μας στην Γεωργία, ασχοληθήκαμε με ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν, με συζητήσεις, ε, απενημερώσεις για την στρατηγική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους αρμόδιους αξιωματικούς και υπαλλήλου. Νομίζω η συζήτηση έγινε με τρόπο επικοδομητικό. Ταξιδέψαμε, μεταφερθήκαμε με ελικόπτερο στην περιοχή Ζουκτίντι, κοντά στα διοικητικά ε, σύνορα, κοντά στην Απχαζία. Προηγουμένως είχαμε επισκεφθεί και την διοικητική γραμμή κοντά στην Τυφλίδα, που, την γραμμή μάλλον που ελέγχεται από το καθεστώς της Τυφλίδας, της Νότιας ω Ε, η επίσκεψη στην Αφχαζία ήταν κάπως πιο δύσκολη να πραγματοποιηθεί, αλλά απευθύναμε ευχαριστίες προς το Κοινοβούλιο της Γεωργίας μας ε, οργάνωσε το ταξίδι αυτό, μας προσέφερε τα μέσα για να ταξιδέψουμε, δηλαδή μας πρόσφερε το ελικόπτερο και μπορέσαμε να δούμε από ψηλά πώς είναι η κατάσταση εκεί. Επισκεφθήκαμε το όρος Ντάμ, το φράγμα ε, που ε, ε, μετά από το έργο υδροελεκτικής ενέργειας παράγει ενέργεια για την περιοχή αυτή, είναι σημαντικό για το εγγύς μέλλον, καθώς και το εργοστάσιο ενέργειας που βρίσκεται κοντά στο φράγμα και που θα πρέπει να ανακαινιστεί και να ε, ανανεωθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτή την ε, υπόθεση. Επίσης, περιπολίες οργανώσαμε στη διοικητική γραμμή που χωρίζει το, την επικράτεια της χώρας από την Αχαζία. Ε, πληροφορηθήκαμε για την ιστορία αυτών των ε, περιοχών και είδαμε σε ποια σημεία είχαν γίνει απαγωγές γεωργιανών. Δυσάρεστες ε, συνθήκες και περιπτώσεις που καταδικάστηκαν από ψηφισμά μας και είναι παράδεκτες. Για την δολοφονία γεωργιανών πολιτών Νομίζω ότι παρουσίασα λίγο πολύ τα όσα συνέβησαν. Εκεί κάποιοι συνάδελφοι από ό,τι κατάλαβα έμειναν παραπάνω στον Πατούμι 10 και 11 Μαΐου συνάντηση της ομάδας φίλων της Γεωργίας. Εγώ χρειάστηκε να επιστρέψω στην Πολωνία Οπότε προείδρευσα σε αυτό το κομμάτι της επίσκεψης μόνο 7 έως 10. Μάλλον ε, έφυγα στο τέλος της 9ης Μαΐου από τη χώρα. Υπήρχαν άλλοι... Αυτά ως προς παρουσίαση. Κύριε Γκάλερ. Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την σύνοψη της επίσκεψης. Πράγματι, έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους Γεωργιανούς. Νομίζω ότι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους από την κορυφή μέχρι τη βάση για να μας εξυπηρετήσουν και η βοήθεια τους φάνηκε χρήσιμη πολλαπλώς. Προσθέσαμε κάποιες συναντήσεις σε πανεπιστήμια όπου ε, μιλήσαμε με φοιτητές στο Βατούμι και στο Τμπιλίσι. Συμμετείχαμε στην ε, Μέρα της Ευρώπης. Πήγαμε και στην Απχαζία, εκτός πόλεων, στην Ήπεθρο. Αξιολογούμε την εφαρμογή της συνθήκη σύμβασης με εισηγητή τον κύριο Μαμίκινς και μετά το καλοκαίρι θα δούμε το θέμα της Γεωργίας με πιο ευρύ και ολοκληρωμένο τρόπο. Οι θέσεις μας ελπίζω ότι θα απηχηθούν και εκεί στην έκθεση αυτή που θα ε, την μετά το καλοκαίρι. ο πρόεδρος ε, της κυβέρνησης παρετήθηκε και είπε ότι θέλει να δώσει στον πρώτο του κόμματός του την ευκαιρία να δημιουργήσει καινούργια κυβέρνηση. Ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός τους λόγω της αλλαγής πρωθυπουργού. Ε, σε λίγο καιρό θα διενεργηθούν και προεδρικές εκλογές. Ε, δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργό παρετήθηκε από μόνος του ή τον εξανάγκασαν σε παρέτηση εξαιτία των διαδηλώσεων που έγιναν. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από το ποιο κυβερνά, εμείς θα είμαστε δίπλα στους Γεωργιανούς. Ευχαριστώ κυρία Μούντι. Δεν απομένουν και πολλά να πω εγώ. Παρ' όλα αυτά κάτι θα πω. Πρώτον, σε σχέση με την αποστολή της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Πιστεύω ότι για μας ήταν πολύ σημαντικό το ότι πήγαμε εκεί και ότι αυτή μας η επισκέψη ε, τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας. Μεταξύ Νότιας Οσετίας και Γεωργίας, όπως είπατε και εσείς, ε, ε, είναι διαπερατά και η κατάσταση εκεί μας ανησυχεί όλους. Μετά την επίσκεψή μας, η κυβέρνηση της Γεωργίας ξεκίνησε το πρόγραμμα «Βήμα για ένα καλύτερο μέλλον», μια ειρνευτική διαδικασία ε, που απευθύνεται στο λαό και στις δύο περιοχές. Ε, έτσι ώστε να επωφεληθούν από τις καλές σχέσεις της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλή αυτή η πρωτοβουλία και πολύ καλό το ότι βρεθήκαμε και εμείς εκεί την εποχή που βρεθήκαμε. Συναντηθήκαμε όπως ε, είπατε και εσείς με πολλούς υψηλούς αξιωματούχους, τον Πρωθυπουργό, υπουργούς, τον πρόεδρο και ήμασταν παρόντες και κάτι διάρκεια του εορτασμού της Μέρας Ευρώπης με ε, ερωτήσεις ε, αρκετά ε, δύσκολες και κρίσιμες που χρειάστηκε να απαντήσουμε προς τους και τους νέους. Όπως είπε ο κ. Γκάλερ, αυτή η επίσκεψη δεν είναι αποκομμένη από τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Είχαμε ένα ψήφισμα την περασμένη εβδομάδα, το οποίο πήρε πολύ δημοσιότητα στη Γεωργία την ίδια από ό,τι έμαθα. Υπογραμμίζει τις καλές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία και τη σημασία της χώρας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος. Ήταν η δεύτερη αποστολή μας κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας μας στη Γεωργία και αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδουμε σε αυτή την χώρα και στην ασφάλεια όλης της περιοχής. Ήταν και μια πολύ πυκνή επίσκεψη με ένα πολύ γεμάτο χρονοδιάγραμμα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σημαντικές συναντήσεις. Στην προηγούμενη μας επίσκεψη την τελευταία είχε γίνει ένας, ένα περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο ενός ανθρώπου και γι' αυτό το λόγο μας ζήτησαν να ε, επισκεφθούμε αυτή τη φορά τα σύνορα. Και στο ψήφισμα μας στηρίξαμε της, ε, την ε, πρόταση για κυρώσεις ε, εν ώψη ε, του περιστατικού οκτωζόρια Νανουκασβίλη. και στις δύο μας επισκέψεις ε, συναντηθήκαμε με ε, πολύ υψηλόβαθμους και ε, εκπροσώπους της ε, στρατιωτικής αποστολής και που κάνουν πολύ καλή δουλειά, πολύ χρήσιμη δουλειά και στηρίζουμε την παράταση θητείας τους εκεί. Ωραία. Τελειώσαμε, οπότε διακόπτουμε για ένα τέταρτο για να περάσουμε μετά στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Θα ξεκινήσουμε ξανά στις 4 με το επόμενο σημείο, το σημείο 13 της ημερησίας διάταξης.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε το επόμενο θέμα στην ημέρησια διάταξη, που, είναι και το τελευταίο ε, σημείο της σημερινής ημέρησιας διάταξης. Τελευταίες εξελίξεις για τις μη στρατιωτικές αποστολές και να σας παρουσιάσω τους ε, διακεκριμένους ομιλητές μας. Δύο τους ξέρετε ήδη πολύ καλά. Γιατί έχουμε συζητήσει την μη στρατιωτική CSDP, τις συγκεκριμένες αποστολές. Έχουμε γνωρίσει ήδη τον κύριο Μπέρτ Φέρμερσεν, που είναι αναπληρωτής, διοικητής για πολιτικές επιχειρήσεις και επικεφαλής αρχηγό του επιτελείου CPCCES, ο κύριο Αγνού Μολενάρ, που είναι υψηλού επίπεδου εμπειρογνώμων στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και τρίτη ε, και εξίσου σημαντική η κυρία Άννα Πένφρατ που είναι ανώτερη αρμόδια πολιτικής του έπλο αποφάσισαν πριν τη συνεδρίαση ότι η εισαγωγή για το θέμα θα γίνει από τον κύριο Μολενάρ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Μπέρτ ε, Φέρσμεσεν και μετά η κυρία Άννα Πένφρατ. Κύριε Μολενάρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ πρόοδος έχει σημειωθεί με βάση την ε, συνολική μας στρατηγική. Η ενίσχυση της πολιτικής ε, πλευράς είναι πολύ σημαντική για το Συμβούλιο και την υπηρεσία μας. Ας θυμηθούμε την κατάσταση τον περασμένο Νοέμβριο. Το Συμβούλιο συμφώνησε για μια διαδικασία με τρεις φάσεις για να ενισχυθεί η μη πολιτική CSDP. Πρώτο καλέσαμε την ε, είπατε εκπρόσωπο να μας παρουσιάσει ένα κείμενο για το μέλλον του πολιτικού CSDP. Δεύτερον, για να υπάρξει ένα <coughs> σχέδιο για την ανάπτυξη της, ε, των δυνατοτήτων του πολιτικού CSDP και κατόπιν η τρίτη φάση θα ήταν να υπάρξει ένα σύμφωνο πολιτικού CSDP για να υπάρξει εφαρμογή. Να δεσμευτούν όλοι ότι θα υπάρξει εφαρμογή. Φέτος Προσπαθήσαμε λοιπόν να εκπονήσουμε αυτό το κείμενο για τη γενική μας ε, προσέγγιση. Το προέτεινε η Πατή Εκπρόσωπος και το ενέκρινε το Συμβούλιο το Μάιο. Η, τα πορίσματα αυτά του Μαΐου είναι πολύ αναλυτικά και λεπτομέρη. Έχουμε τους εξής στόχους. Πρώτον, ενίσχυση της αποτελεσματικότητα της πολιτικής ΙΣΤΠ και των αποστολών τη και να ενισχύσουμε τη δυνατότητα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των ε, προκλήσεων. Καλό σημείο αφετηρίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 10 αποστολές και έχουμε πολύ πείρα που μας επιτρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Για παράδειγμα, για να ανταποκρινόμεθα συντόμως. Ο συνάδελφός μου, ο Μπέρτ, θα πει περισσότερα γι' αυτό. Ένα άλλο βασικό στοιχείο της δουλειάς μας. Η ασφάλεια της Ευρώπης ξεκινάει πέρα από τα όρια μας και οι αποστολές ε, αυτές μπορούν να βοηθήσουν να προστατεύσουμε και τη δική μας ασφάλεια. Αυτό δεν είναι τελείως ε, νέο, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι περισσότερες δυνατότητε για, πολιτική, για αποστολές της ε, πολιτικής CSDP, αστυνομικοί, δικαστές, άλλοι προγνώμονες, βεβαίως ε, είναι σε μεγάλη ζήτηση και στο εσωτερικό της Ένωσης. Αυτό λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο προσεγγίζουμε το θέμα γενικά, αλλά τώρα που περάσαμε και στην ε, ανάπτυξη των ε, δυνατοτήτων. Σας διαβεβαιώ ότι το νομικό πλαίσιο του CSDP δεν έχει αλλάξει, τα άρθρα της ηθίκης δηλαδή, και η, ο καθορισμός της εντολής θα γίνεται με τις ίδιες διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι οι προτεραιότητές μας που ήταν η αστυνομία, το κράτος δικαίου και η δημόσια δίκηση θα εξακολουθήσουν να είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Η CSDP προσπαθεί να αντιμετωπίσει κρίσεις ή σειράξεις. Το σημείο φετηρίας είναι κοινή ανάλυση της κατάστασης και έχουμε προτείνει το PFCA, το πολιτικό πλαίσιο για την ε, προσέγγιση των κρίσεων. Είναι μια ολιστική ανάλυση του περιβάλλοντος το οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε. Και πώς θα πρέπει να ανταποκριθεί η Και μέσω της CSDP. Εάν αποφασίσουμε να ε, υπάρξει αποστολή, θα το κάνουμε αναλύοντας επιτόπου τη συγκεκριμένη κατάσταση με βάση την ολοκληρωμένη προσέγγιση για να υπάρξει και συνεργασία με άλλα προγράμματα της Κομισιόν. Και αυτό νομίζω πως ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη. Στο κείμενο αυτό το θεωρητικό που παρουσίασε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος τον Απρίλιο αποφασίσαμε στο μέλλον οι αποστολές μας να είναι πιο ε, ε και να μπορούν να αναπτύσσονται ή να μειώνονται σε ε, διαστάσεις ταχύτατα να είναι κλιμακόσμες και αποκλιμακόσμες. Αυτό ε, βεβαίως θα το δούμε ε, στο μέσο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Και θα έχουμε και ποσοτικούς δείκτες για να σημειώσουμε την πρόοδο ή την έλλειψη πρόοδου προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να μπορέσουμε να επανεστιάσουμε αν χρειαστεί. Αυτή λοιπόν η κλιμακωτή προσέγγιση είναι η βάση του κειμένου μας. Για να καθορίσουμε τι θα περιείχε η εντολή μιας αποστολή για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένε προκλήσει ασφάλεια, φυσικά ανάλογα με τι καταστάσει. Επίση, σημειώνω ότι έχουμε ήδη πρότυπα από τι ε, ενεξελίξει αποστολέ που αντιμετωπίζουν ε, τα θέματα μετανάστευση, έλεγχο των συνόρων, τρομοκρατία κτλ. Κέντρο όλα αυτά είναι η ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ της ESDP και άλλων για να αντιμετωπίσουμε και τους ε, κινδύνους στο εσωτερικό και ευρύτερα. Πρέπει να συμμετέχουν ε, στην ε, διαμόρφωση των προγραμμάτων μας και άλλοι φορείς όπως η Frontex. Αυτά πρέπει να τα δούμε πιο συστηματικά και να βοηθήσουν και οι κυβερνήσει διαφόρων κρατών μελών, καθώ και οι προπαρασκευαστικέ ομάδε προπαρασκευαστικές ομάδες του Συμβουλίου. Η ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ τη SDP και το JJ ε, θα μας βοηθήσει. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, ορισμένες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας που τη χρησιμοποιούν και για τους στόχους της e Άρα πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε την πιο λογική προσέγγιση. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η ανάπτυξη, η εκπόνηση αυτού του προγράμματος για την πολιτική CSDP. Είναι εν εξελίξη. Αναλύουμε τις ανάγκες που προκύπτουν από τους στρατηγικούς μας στόχους και θέλουμε να εισαγάγουμε και μεθόδους για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητε. Για παράδειγμα, εκπαίδευση και κατάρτιση, οργανωτικά μέτρα, αλλά και κίνητρα για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα. Θέλουμε μέχρι το καλοκαίρι τρέχοντος, δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες, να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό θα μας βοηθήσει κατόπιν να καταλήξουμε σε αυτό το σύμφωνο για το CSTP που θα πρέπει να συμφωνηθεί μέχρι τον Νοέμβριο τρέχοντος. Η ουσία αυτού του συμφώνου θα είναι να δεσμευθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να υπάρξουν οι αναγκαίες βελτιώσεις για να ενισχυθεί η πολιτική CSDP και από πλευράς προγραμματισμού και από πλευράς ανάπτυξης δυνατοτήτων. Η Επιτροπή και η Υπηρεσία εξωτερική Δράσης θα μας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία και θα μας στηρίξουν. Νομίζω λοιπόν ότι καλά έχουμε ξεκινήσει, αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή. Και είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη για να επιτύχουμε τα επιτυχόμενα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μόλνερ. Τώρα ο λόγος στον κύριο Μπέρτ Βέσμερσεν. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο επιχειρησιακό επίπεδο θα ήθελα να αναπτύξω κάποια ζητήματα που ίσως να είναι τεχνικότερα, αλλά θα ζητήσω την υπομονή σας. Όπως είπε ο κύριος Μολνάτ, έχουμε μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε. Με 200.000 άτομα και μια πολύ καλή επισκόπηση από τις 15 Μαΐου για τις 10 επιχειρήσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής μας πρέπει να δούμε πώς αυτές οι αποστολές μπορούν να περάσουν στην οικοδόμηση δυνατοτήτων πέρα από την διαχείριση κρίσεων και να διασφαλίσουν να προστατεύσουν την Ευρώπη και τους πολίτες της. Στα σχόλιά μου θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό που έχουμε ονομάσει την κλιμακωτή προσέγγιση, την ε, δυνατότητα απόκρισης και το λεγόμενο warehouse, το πλωστάσιο εδώ για τη γρήγορη ανάπτυξη δυνάμεων. Είναι πολλά τα στοιχεία που επηρεάζουν τη γρήγορη ανάπτυξη των δυνάμεων. Δεν υπάρχει βεβαίω εδώ τέλεια λύση και ένα βασικό στοιχείο είναι το πόσο γρήγορα λαμβάνονται αποφάσει που δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε εμεί. Το μίσο που ελέγχουμε λίγο περισσότερα τα πράγματα είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων, η ενδεχόμενη ανάπτυξη ε, προσωπικού ή στρατιωτικού προσωπικού ε, σε εφεδρεία Πρέπει να αυξήσουμε την ικανότητα της Ένωσης να επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την εντολή της μόλις ληφθεί μια απόφαση. Αυτό είναι το θέμα για μας βέβαια, να λαμβάνεται μια απόφαση. Τότε να μπορούμε να αναπτύξουμε το... να στείλουμε το στράτευμα και να αναλάβει δράση επιτόπου. Τι ονομάζουμε τώρα πολυεπίπεδη κλιμακωτή προσέγγιση. Τρία επίπεδα περιλαμβάνει. Αυτό που ονομάζουμε τη δυνατότητα απόκρισης. Μετά τους πόρους των κρατών μελών, αυτούς που έχουν συνενωθεί βάσει μιας γρήγορης πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και μετά μια διαδικασία για επιχείρηση. Αυτή την πολυεπίπεδη διαδικασία την ε, εκτελούμε βάσει, της, βάσει εργαλείων και μέσων από προπαρασκευαστικές δράσεις, ανταλλαγή προσωπικού, δεν θα περάσω τώρα σε λεπτομέρειες. Ε, η πρώτη φάση, το πρώτο επίπεδο είναι ζωτική σημασία. Αφού ληφθεί μια απόφαση, ελπίζαμε να έχουμε ένα αριθμό ε, ανθρώπων που μπορούμε να αποστείλουμε να αναπτύξουμε γρήγορα. Έτσι λειτουργεί ο ΙΕ, ας πούμε σε περιπτώσεις και πολιτική και ιστορικής προστασία. Αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και την απόφασή του το 2017. Δεν υπάρχει τέτοιο σώμα ακόμα. Όμως έχουμε 30 ανθρώπους στην ε, ε, δυνατότητα απόκριση, εκ των οποίων 22 συμμετέχουν στι αποστολέ. Αυτή τη στιγμή είναι απεσταλμένοι εκεί που πρέπει και ενημερώνουν την πλατφόρμα για τις αποστολές εδώ στις Βρυξέλλες. Αυτό το πλάνο έχει ήδη εγκριθεί και η δυνατότητα απόκρισης ήδη λειτουργεί. Άρα έχουμε 22 συγκεκριμένους υπαλλήλου που ήδη έχουν αναλάβει δράση στις ε, διάφορες αυτές επιχειρήσεις και αποτελούν μέρος της ομάδας για τη δυνατότητα απόκρισης. Έχουν γενικές γνώσεις, στοιχεία που πάντα χρειαζόμαστε, όπως ασφάλεια, προμήθειες, ανθρώπινη πόροι, έχουν λοιπόν γενικέ γνώσει ούτω ή άλλω, τα χρειαζόμαστε αυτά, αλλά και ειδικότερε. Αυτέ ε, εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη εντολή κάθε φορά. Το άλλο στοιχείο είναι η ενισχυμένη πλατφόρμα αποστολών. Η διοικητική επιμελητία, η CIS, οι προμήθειες είναι πράγματα που καλύπτονται σε αυτή τη πλατφόρμα. Όταν το Συμβούλιο λοιπόν αποφασίζει μια απόσταση, αποστολή, μπορούμε γρήγορα να αποστείλουμε κάποιον στην περιοχή τη αποστολή, στην έναρξη τη. Άλλε αρμοδιότητε των ανθρώπων αυτών μπορεί να είναι επικουρικό, να χρησιμοποιήσουν, να αναλάβουν κάποια άλλη δράση, όπως κάποιο λιμάνι, ε, όπως κάτι πολύ συγκεκριμένο σε κάποιο λιμάνι σε μια ξένη χώρα. Ε, έξι εβδομάδες χρειάζεται η διοργάνωση της ομάδας που εξυπηρετούν και άλλες ειδικέ ομάδες από τα κράτη-μέλη ή άλλοι ειδικοί σχηματισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Χωροφυλακή. Αυτή η δυνατότητα απόκρισης υποστηρίζει την άλλη δύναμη που κανονικά θα θέλαμε να αποστείλουμε και που μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο να αποσταλεί. Τώρα, για την ε, EU-UN iraq τη συγκεκριμένη αυτή αποστολή. Δανειστήκαμε κόσμο από άλλες αποστολές για να την επαντρώσουμε. Και αυτό επειδή είχαμε απόφαση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο και ανάπτυξη ήδη τον Νοέμβριο. Ο κατάλογος έχει ήδη καταρτιστεί, οπότε φαίνεται ότι εδώ η δυνατότητα ε, εκτύπλωσης λειτουργήσε αποτελεσματικά. Δεν θα πρέπει όμως εδώ να προσπαθούμε με τα μέσα του ενός να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ε, δηλαδή, το δάνειο από αλληλεποστολή μπορούσε να γίνει για ένα δεκαπενθήμερο μόνο. Θα πρέπει να βρεθεί μια ε, διαρκέστερη λύση και αυτό εξαρτάται από την πολιτική εντολή που θα λάβουν οι επιχειρήσεις. Τώρα ως προς την αποθήκη, το πλωστάσιο αυτό, μια άλλη πρόσφατη εξέλιξη, ε, ο εξοπλισμός είναι σημαντικός σε οποιαδήποτε γρήγορη ε, αποστολή. Μπορούμε να στείλουμε ειδικού, αλλά χωρίς κανένα εξοπλισμό, στρατιωτικό, ε, φαρμακευτικό, ιατρικό, δεν μπορούν να προσφέρουν και πολλά. Είναι μονόδρομος λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλωστάσιο για την υποστήριξη νέων αποστολών μόνο όμως. Διότι έτσι κι αλλιώ ο εξοπλισμό καθίσταται απειρχαιωμένο πολύ γρήγορα. Έχουμε υπογράψει συμβάσει πριν από τρεις εβδομάδε μόλις για το νέο αυτό οπλοστάσιο ή αποθήκη το οποίο εγκαινιάστηκε στην Σουηδία με σκοπό να αποθηκεύεται εκεί βασικός εξοπλισμός για τη γρήγορη εκδήλωση των αποστολών και για να έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε την αποστολή νέων αποστολών με 200 ε, ανθρώπους σε 30 μέρες. Έτσι, ο εξοπλισμός μεταξύ των αποστολών αποστέλλεται εξορθολογισμένα Και αυτό για τις επιχειρήσεις του άρθρου 20 και τους ειδικού απεσταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 610 οχήματα, 2.000 υπολογιστές, 600 λάπτοπ, είναι μέρη του εξοπλισμού, του ζωντανού αυτού υλικού που θα περιλαμβάνει η αποθήκη, το πλωστάσιο. Επίσης κάποιες υπηρεσίε που θα χορηγούνται σκοπεύουν να αυξήσουν την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την σωστή χρήση των υπαρχόντων πόρων μας. Μια κεντρική βάση δεδομένων επίσης και ό,τι πλεόνασμα μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλους πόρους. Είναι σημαντικό αυτό από χειρισιακής σκοπιάς. όχι μόνο για τη διαδικασία υποβολής, ενδιαφέροντος μπορεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα, αλλά για να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα. Ένα άλλο θέμα είναι η διαλειτουργικότητα, διότι έχουμε προσωπικό που μετακινείται μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών και περνάει από τη μια αποστολή στην άλλη, οπότε πρέπει να γνωρίζουν καλά τον εξοπλισμό μα. Θα ολοκληρώσω εδώ, Πρόεδρε, και με συγχωρείτε που ήμουν κάπω πιο τεχνικό, αλλά όσο πιο χειροπιαστά πράγματα ε, αναπτύσσει κανεί, τόσο πιο τεχνικά γίνονται. Ελπίζουμε οι δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, αποστέλλονται επί τόπου πολύ πιο γρήγορα και στα πρώτα στάδια μια αποστολή είναι πολύ σημαντικό το πώ εκδιπλώνεται αυτή για λόγου αξιοπιστία. Πράγμα που είδαμε στην αποστολή μα στο Ιράκ, α πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Με την εμπειρία μας από τις επισκέψεις μας έχουμε κατανοήσει τα προβλήματα που έχουν σχέση με τεχνικά ζητήματα, με εξοπλισμό και με την ανάπτυξη των κατάλληλων μονάδων μας. Χρειάζεται να ενοποιήσουμε και να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε τις μεθόδους μας, τη μεθοδολογία μας για να γίνουν οι αποστολές μας πιο αποτελεσματικές. Thank Η κυρία Άννα Εργάζομαι για την ε, EPLO με 37 μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, που ασχολούνται με θέματα ειρήνευσης. Ε, εμείς είμαστε ένας ενδιάμεσος, liaison office όπως λέμε, και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε τη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, πώς μπορεί η Κομισιόν να βοηθήσει σε μια, στην ανάπτυξη μιας βιώσιμας, βιώσιμης ειρήνης. Ε, τέρους εντάσσοντας ε, μια διάσταση ασφάλειας των μεμονωμένων ατόμων ε, στη δράση μας, όχι μόνο της ασφάλειας του κράτους γενικότερα ή των ε, επισήμων. Γι' αυτό το λόγο διοργανώνουμε τακτικά φόρουμ διαλόγου προκειμένου όλες οι προοπτικές ασφάλειες να λαμβάνονται υπόψη εξίσου στη δράση μας. Εξετάζοντας τις εξελίξεις εν ώψη του συμφώνου, ε, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα έχουν συμβεί ήδη, αλλά έχουμε και πολλές προκλήσεις και κινδύνους για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση με την υιοθέτηση του ίδιου του συμφώνου. Θετικές εξελίξεις. η εξής στα συμπεράσματα του Συμβουλίου αλλά και στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις είδαμε ότι δίνεται η ευκαιρία πλέον οι, οι αποστολές μας, οι αποστολές της ε, CSTP να χρησιμεύσουν και για την εδραίωση μιας ε, βιώσιμης ειρήνης. δίνεται επίσης έμφαση στην αποκοινού ανάλυση. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό δεν το ξέρουμε πολύ καλά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ανάλυση που θα γίνεται κάθε φορά της, ε, ε της σύγκρουσης ε, είναι αρκετά ελκυστική έτσι ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Σε πολλά έγγραφα, ιδιαίτερα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ε, γίνεται λόγος για την συμμετοχή ε, και τη συνειδητοποίηση των ε, επιτόπιων εμπλεκόμενων παραγόντων. Και επίσης γίνεται λόγος για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση έχοντας στο μυαλό μας πώς μπορούμε να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτηματικά για το πώς όλα αυτά θα αναπτυχθούν σε επόμενους μήνες, αλλά πριν από αυτό να ε, υπογραμμίσω την εξής πρόκληση. Η ισορροπία ανάμεσα στην βραχυπρόθεσμη ασφάλεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της χώρας στην οποία δρούμε. Οι ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανάγκη προφανώς να δείχνουν ότι πετυχαίνουν στόχους γρήγορα. Αλλά πολλές φορές το βραχυπρόθεσμο δεν είναι συμβατό με το μακροπρόθεσμο. Μερικές φορές μπορεί να γίνει, μερικές φορές όχι. Σε στρατηγικό επίπεδο, όταν ξεκινάμε μια αποστολή, μπορούμε να δικαιολογήσουμε σε ένα βαθμό ότι, το, ότι γίνεται για να εξασφαλιστούν τα βαραχυπρόθεσμα εσωτερικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, πέραν των άμεσων απειλών για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπιστούν, πρέπει πάντοτε να βλέπουμε και πιο μακριά. Πώς η αποστολή μας πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλλει μακροπρόθεσμα για την, στην ειρήνη της περιοχής στην οποία επιχειρούμε. Ε, ποιους θα υποστηρίξουμε, πού ακριβώς θα αναπτύξουμε την αποστολή μας και ποιος είναι ο στόχος μας, ε, ο τελικός μας στόχος και πώς μπορεί να μετρηθεί τι θα θεωρηθεί επιτυχία τελικά. Αν αυτά δεν τα έχουμε στο μυαλό μας από την αρχή, τότε μπορεί η δική μας παρέμβαση μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να βλάψει την ασφάλεια της χώρας στην οποία επιχειρούμε. Πρέπει να ξέρουμε πώς θέλουμε να επηρεάσουμε την δυναμική της ε, σύραξη στην οποία παρεμβαίνουμε. Η UNDP έχει στοιχεία για το πώς μερικές φορές η αντιτρομοκρατική δράση μπορεί να πυροδοτήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Επίσης, οργανωμένο έγκλημα στην Μεσόγειο. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο τη λαθρομετανάστευση και όχι την λαθρέα, ε, το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Ε, στη χειρότερη περίπτωση, λαμβάνοντα υπόψη μόνο τη μετανάστευση, μπορεί να είμαστε πραγματικά πολύ αντιπαραγωγικοί. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε και τι προτεραιότητε των κρατών μελών, αλλά και την πιο μακρο, το πιο μακροπρόθεσμο όραμα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ονομάζουμε local ownership. Τι εννοώ, είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την άποψη ε, των διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού. Είναι σημαντικό αυτό προκειμένου πραγματικά να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα, τα αληθινά προβλήματα. Επίσης, πρέπει να επενδύσουμε σε μια σωστή ανάλυση. Αυτή η ανάλυση δεν πρέπει να γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής, αλλά και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ε, και της για τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης. Γιατί θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθούμε το πώς η επιχείρησή μας επηρεάζει την πραγματική δυναμική της σύραξης. Επιδραθετικά ή βλάπτη. Και όταν χρειάζεται να προσαρμόζουμε τις, ε, τη δράση μας το ονομάζουμε conflict sensitivity, δηλαδή ευαισθησία έναντι της επίδρασης που έχουμε εμείς στην ίδια τη σύραξη. Μόνο αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των σειράξεων. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει. Πολλά έχουν σχέση με το σύνδεσμο μεταξύ Jai και αποστολών CSTP. Αφενός διότι ε, ανταγωνίζεται για τους ίδιους πόρους, αλλά απ' την άλλη και αφετέρου γιατί οι αποστολέ ΚΠΕ, ε, ΚΠΑ, συγγνώμη, ε, μπορούν να ε, επηρεάσουν με διάφορους τρόπους την κατάσταση επιτόπου ε, Λαμβάνοντα όμως υπόψη τη γνώμη πολλών διαφορετικών εμπειρογνωμόνων. Οπότε δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στη συνεργασία με τον τομέα της δικαιοσύνης και της εσωτερικής ασφάλειας. Σε συνεργασία βέβαια με αυτούς θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν και αυτή την ίδια ευαισθησία έναντι των αποτελεσμάτων της δράσης τους. Γιατί αυτοί δεν έχουν τόση πολλή εμπειρία σε δράση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να τους διδάξουμε. Και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους φορείς του Τζάι, του πυλώνα δικαιοσύνης εσωτερικών υποθέσεων, να κινητοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να εντάξουμε αυτή την έννοια της ευαισθησίας ε, και στο σύμφωνο όταν το αναπτύξουμε. Οι εμπειρογνώμονες παρακολούθησης και αξιολόγησης θα πρέπει να ενταχθούν ε, στις ε, προϋποθέσεις πόρων και δυναμικού που θα πρέπει να τσεκάρουμε ότι έχουμε πριν ξεκινάμε οποιαδήποτε επιχείρηση. Και προφανώς να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη και στην εκπαίδευση εκείμνας που γίνεται πριν από την επιχείρηση, ε, στην περιγραφή των θέσεων εργασίας τις οποίες θα προκηρύξουμε, για τις οποίες θα ζητήσουμε προσωπικό, ε, έτσι ώστε να ξέρουμε εκ των προτέρων σε τι θέλουμε να συνεισφέρουμε. Τέλος, για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο με το πολιτικό βάρος που έχει θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ασφάλεια των μεμονωμένων ατόμων του πληθυσμού ε, έτσι ώστε πραγματικά οι αποστολές μας να οδηγούν σε μείωση της βίας και αύξηση των πιθανότητων βιώσιμης ειρήνης. Και ΠΑΑ δεν είναι ένα μακροπρόθεσμο εργαλείο, αλλά ως βραχυπρόθεσμο εργαλείο θα πρέπει να συνεισφέρει στη μακροπνοηρήνη. Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συνεχίσει να πιέζει τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ε, προβαίνουν σε συνεχή αξιολόγηση της δράσης μας και να εντάξουν την ευαισθησία ε, στην ε, δράση τους. Ε, τα ίδια θέματα μπορείτε να θίγετε και όταν έχετε επισκέπτες, εξωτερικούς επισκέπτες, ε, πυρογνώμονες ή πολιτικούς από ξένες χώρες. Μπορείτε αυτό να το οργανώσετε στο πλαίσιο συνεδρίων ανοιχτών, στο πλαίσιο κλειστών συναντήσεων. Επίσης, ο το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, προασπίσει τον προπολογισμό της ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Πώ μπορεί αυτό ο προπολογισμό να χρησιμοποιηθεί πιο σωστά και να διατηρηθεί. Τελειώνοντας, επαναλαμβάνω γιατί θεωρώ πως είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην ασφάλεια των ατόμων στις ε, χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πρώτον, γιατί αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, αλλά και δεύτερον, για να γίνει πιο αποτελεσματική η δράση μας. Γιατί αν δεν εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσκάπτουμε και το δικό μας μέλλον. Η μη στρατιωτική και πρέπει να δώσει το παράδειγμα, έτσι ώστε οι συζητήσεις να ξεκινήσουν και με την στρατιωτική και Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει το λόγο κύριε Μποστινάρου. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά ήρθα πολύ αργά γιατί είχα πολλές άλλες υποχρεώσεις. Με συγχωρείτε. Δεν θα πάρω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τότε να κάνω εγώ ερωτήσεις. που απευθύνεται σε όλους και στους τρεις σας. Σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχουν ε, πολλοί φορείς. Για παράδειγμα έχουμε σε μια περιοχή μια πολιτική αποστολή της Ένωσης μια λίγο διαφορετική αποστολή του ΝΑΤΟ και επίσης ε, αποστολές κάποιων κρατών μελών. για να αντιμετωπίσουμε σειρά προβλημάτων σε μια χώρα που είναι σε αναβρασμό. με πολλούς ακραίους ε, να δρουν. Τι εννοείται επιμέτρου αποστολές. Δεν υπάρχει ανάγκη να συντονιστούν οι διάφοροι που θα αποφασίσουν πώς ακριβώς θα κοπεί το ύφασμα για αυτήν την επιμέτρου αποστολή. Πώς θέλετε να απαντήσετε με τη σειρά που είναι αρχικές ομιλίες αρχικέ ομιλίε ή πώς θέλετε. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Ένα θέμα που μας απασχολεί συχνά, όπου υπάρχει κάποια σύραξη, συμμετέχουν διάφοροι. Κάποιοι ήδη έχουν εμπλακεί, μετά έρχεται CSDP, ή μετά ε, από την CSDP μπορεί να έρθει μια στρατιωτική αποστολή ή πριν και κάθε κατάσταση είναι βέβαια διαφορετική. Γι' αυτό τόνισα ότι πρέπει να γίνει εκ των προτέρων μια κοινή ανάλυση με την DEVCO, με την GHA, με την Επιτροπή, με την EAS, με τους πολιτικούς σχεδιαστέ, τους στρατιωτικού σχεδιαστέ, για να έχουμε μια καλή επισκόπηση της κατάστασης, να αναλύσουμε τη δυναμική της σύγκρουσης, να λάβουμε υπόψη όλες τις πλευρέ. να δούμε πώς συνδέονται τα θέματα, ποιοι είναι κύριοι πέτοι για την κρίση και τη σύγκρουση, πώς λοιπόν να προσαρμόσουμε την δράση μα. αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία της ε, ολοκληρωμένης προσέγγισης. από το σχεδιασμό της επιχείρησης μέχρι και την δράση επιτόπου για να υπάρξει συντονισμένη δράση. Θαυμάσια και η παρέμβαση της συναδέλφου μου εδώ. Το βασικό είναι επίσης να ε, πιστεί ο τοπικός πληθυσμός για τη σκοπιμότητα αυτών που κάνουμε. Βεβαίω οι αποφάσει λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη εδώ στι Βρυξέλλε, από το Συμβούλιο. Αλλά η ανάλυση πρέπει να είναι όσο πληρέστερη γίνεται. Και τα κράτη-μέλη έχουν ε, και τις δικές τους πηγές πληροφόρησης και αντένες στα κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η αποστολή σε σχέση με την εξελισσόμενη κατάσταση Βέβαια οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα κράτη-μέλη. Άρα πρέπει να τους δώσουμε τη σωστή πληροφόρηση. Αλλά δική τους απόφαση είναι. Μπορεί να πούν ε, δεν προχωράει η αποστολή αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, ενεργούμε, να επιχειρούμε εκεί ή αλλιώ να πούνε όχι, τα μαζεύουμε. Συνολικά, όπως σωστά είπατε κι εσείς, πρέπει να συνδυάσουμε όλες τις συνιστώσεις της προσπάθειάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για παράδειγμα, να δούμε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Το Μαλί είναι παρόντα τα Ηνωμένα Έθνη με στρατιωτική και πολιτική αποστολή. Υπάρχουν εθνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Διάφοροι εμπλέκονται. Ορισμένοι χρηματοδοτούν ε, επιτόπου προγράμματα και το τι θα κάνουν και οι άλλοι βεσκά μας ενδιαφέρει και εμάς όταν εμείς προγραμματίζουμε. Σε κάθε έγγραφο σχεδιασμού πάντα υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει αυτό κάνουν οι άλλοι που συμμετέχουν άρα δεν θα μπούμε στα χωράφια τους. Σε πολλές αποστολές ο συντονισμός είναι βασικό μέλημά μας. Και πάλι στο Μαλή να αναφερθώ η Κομισιόν. Προωθεί το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων από την τοπική κυβέρνηση. Και βέβαια θα έπρεπε και η κυβέρνηση του Μαλή. Αυτό θα ήταν το ιδεώδες. Η κυβέρνηση του Μαλή να συντονίζει τις προσπάθειες όλων των ε, παρεμβαινόντων Αλλά δεν έχουν δυνατότητα δυστυχώς. Υπάρχει πολλή δουλειά, όλοι οι Γαλλοί μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί η κατάσταση είναι συνήθως δεινή. Ιράκ, τελευταία μας αποστολή. Όταν την προγραμματίζαμε, βέβαια μελετήσαμε τι έκανε το ΝΑΤΟ που ήταν παρόν και κάποια κράτη-μέλη, τι έκαναν τα Ηνωμένα Έθνη για την ασφάλεια και το ΝΑΤΟ προτίθεται τώρα να αυξήσει την παρουσία του εκεί. Ουσιοδό. Και εκεί έχουμε πολύ τακτικέ επαφές για να αλληλοσυλλογωνόμεθα και να μην ε, μπερδευόμαστε. Εμείς ασχολούμαστε κυρίως με την πολιτική πλευρά. Εργαζόμαστε με τον Σύμβουλο ε, Εθνικής Ασφαλείας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τώρα η κυρία Αναπενφρά. Ναι. Υπάρχουν πολλοί εμπλεκομένοι παράγοντες εδώ, πολιτικοί και στρατιωτικοί. Και πρέπει πάντοτε να διερωτόμαστε ποια είναι η προστιθέμενη αξία σε κάθε περίπτωση. Τα κράτη-μέλη μπορεί να αποφασίσουν να οργανώσουν μια αποστολή για διαφορετικού λόγους σε κάθε περίπτωση. Απλώς θα έλεγα όταν γίνεται αυτό το χαρτογράφηση, το οργανόγραμμα, ποιο κάνει τι, είναι το θέμα να δούμε και τι κάνουν οι διάφορες ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνία των πολιτών. Πολλές φορές έχουν και αυτοί ε, κάποιες ε, πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές, όπως η οικοδόμηση δυνατοτήτων και βοηθούν στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, στατικών δυνάμεων και του τοπικού πληθυσμού. Μια από τι προστιθέμενε αξίε των δικών μας αποστολών σε αυτήν την ε, περίπτωση είναι να ενισχύουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης και να επιτρέπουμε στις δυνάμεις ασφαλείας να προβάλλουν τη δυνατότητα να σταθεροποιήσουν την κατάσταση για τον τοπικό πληθυσμό. Αυτά. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι απαντήθηκαν οι ερωτήσεις και εξαντλήθηκε ο κατάλογος ομιλητών σε αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό μια άλλη φορά. Κατά πάσα πιθανότητα ε, προσκαλώντας επικεφαλής των ίδιων των επιχειρήσεων. Σε κάποιο βαθμό υπήρξαν κάποια προβλήματα πριν από λίγο καιρό. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί και επιπλέον μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση επιτόπου. επισκεπτόμενοι μια σειρά από επιχειρήσει σε μια σειρά από περιοχέ. Και εμεί συγκεντρώνουμε χρήσιμε εμπειρίε, βλέποντας αυτή την ποικιλία διαφορετικών περιπτώσεων. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα μας λείπει είναι μια συνολική εικόνα του τι συμβαίνει με την κοινωνία των πολιτών. Από καιρού εις καιρών Πρέπει να συναντιόμαστε, προσπαθούμε να συναντιόμαστε για να συνδυάσουμε αυτού του είδους τις επιτόπιες συναντήσεις με εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, όχι, μάλλον ε, είναι από τις λίγες φορές που δεν είναι εύκολο να έχουμε επιτυχία για να το συγκεντρώσουμε όλους ταυτόχρονα στο ίδιο μέρος και να βρούμε και τα κατάλληλα χρονικά σημεία που να είναι διαθέσιμα και οι Δεν είναι πολύ απλό. Αλλά ναι, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ενδυναμώσουμε αυτές τις δυνατότητες. Όποτε μπορούμε να κάνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, είναι προφανές ότι θα το κάνουμε. Πολύ σας ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, διάφορα. Δεν ε, βλέπω να υπάρχει κάτι. Σας θυμίζω ότι η ερχόμενη συνεδρία είναι στις 11 Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ. I would like to, to... Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς οι οποίοι ήταν πολύ απασχολημένοι σήμερα και την γραμματεία. Ευχαριστούμε. <laughs>